Pan Preda. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, denní zasedání. το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξή μας είναι το, η έκθεση της κυρίας Μπαλσάνη σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 1 κάθετος 2012 χρηματοδότηση του προγράμματος ΙΤΕΡ. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπαλσάνη αμέσως. Grazie Presidente. Eh, cari colleghi, carissimo Commissario,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 Αγαπητή Φρανσέσκα, εκ μέρους της Κομισιόν, χαίρομαι για την υποβολή της έκθεσής σας και χαίρομαι και για τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία 1η Δεκεμβρίου πέρυσι για πρόσθετη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ για κατά 1,3 δις για το 2012 και 2013. Αυτός σημαίνει ότι 100 ήδη περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό του 2012 και αυξάνουμε τις οροφές για φέτος το 2 και στο 5 και βεβαίως δεν προκρίνουμε την εφαρμογή και τι πρέπει να γίνει για το 2013 διότι άλλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στις διαπραγματεύσεις για τον ε, προϋπολογισμό του επόμενου έτους είναι που να βρούμε ακόμη 360 εκατομμύρια χωρίς να βλάψουμε οποιαδήποτε από τα άλλα σχέδια για την καινοτόμο και ανταγωνιστική Ευρώπη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Δύο λεπτά ο κύριος Λαβία πρώτος. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπω τόνισε η συνάδελφο Μπαλτσάνη, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 1 του 2012 αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη διοργανικά με την ευκαιρία τη περάτωση διαδικασία του προπολογισμού του 2012 με τη χρηματοδότηση 1,3 ε, ε, εκατομμυρίων ευρώ πρόσθετου κόστου για το ΙΤΕΡ για την περίοδο 12-13. Συγκεκριμένη περίπτωση, το σχέδιο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού προβλέπει την αύξηση κατά 650 εκατομμύρια ευρώ για το κεφάλαιο 1α για το 2012. Υποστηρίζουμε την έκθεση τη κυρία Μπαλτσάνη και ζητάμε κατά συνέπεια να δοθεί θετική ψήφο για να τιμηθεί η συμφωνία που επετέφθη μεταξύ των δύο αρχών του προπολογισμού με τη διαμεσολάβηση τη Επιτροπή στο τέλο τη προηγούμενη χρονιά. Εκμεταλλεύουμε την ευκαιρία αυτή για να θυμίσω ότι το σχέδιο ή το πρόγραμμα ITER θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που θα ζητήσουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και που θα οδηγήσουν στην έγκριση του προπολογισμού για το 2013. Διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν σύντομα εν ώψη της, ε, δημοσίευση του σχεδίου προπολογισμού που θα υποβληθεί στι 25 ε, Απριλίου από τον Επιτρόπο Λεπαντόφσκι. όπω ήδη αναφέρθηκε στι κατευθυντηρίου γραμμέ του προπολογισμού που ενεκρίθη από το Κοινοβούλιο αυτό, περιμένουμε 460 εκατομμύρια ευρώ που έχουν συμφωνηθεί για τη χρηματοδότηση του επιπρόσθετου κόστου του, του προγράμματος ΣΥΤΕΡ που θα αφορούν τον προπολογισμό του 2013 θα ε, Μα τα εγγυηθούν δίχως αυτό να έχει επίπτωση σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στι πολιτικές που συμβάνουν στην επίτευξη των στόχων της, Ευρωπαϊ... της ε, ε, Ευρώπη. Ε, αναφέραμε ότι αυτές είναι οι στρατηγικές μας προτεραιότητες, οι οποίες βρίσκουν σύμφωνο, σύμφωνο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, η κυρία Χέρτσοκ για 3,5 λεπτά τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, εν ονόματι της σοσιαλιστικής ομάδος χαιρετίζω την έκθεση αυτή και χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μεγάλες ε, πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σκέφτονται προς την ίδια κατεύθυνση και θα μπορέσουμε να αναδιοργανώσουμε την διάθεση των πόρων μας κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να καθησυχαστούμε. Πρέπει να προσθέσουμε ότι η αύξηση των πόρων θα μπορέσει να καλέψει σημεία του προϋπολογισμού που είχαν καθυστερήσει λόγω ασαφίας και αυτή η καθυστέρηση θα δημιουργήσει αύξηση του κόστους και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο για την περίοδο 2012-2013 αλλά μέχρι και το 2020. Εξού και είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διακηρύξουν την πολιτική θέλησή τους και την επιθυμία τους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή κατά τρόπον ώστε τα, οι τάσεις στα θέματα της ενεργείας και της παγκοσμιοποίησης να μπορέσουν να προωθηθούν και οι νέες ομάδες συμφερόντων που εμφανίζονται στον τομέα της ενεργείας που είναι τώρα ε, πιο μεγάλα συμφέροντα από ό,τι στο παρελθόν να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θυμηθεί πότε ξεκινήσαμε το πρόγραμμα τέρ μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τότε ο Κορβατσόφ που ήταν γενικός γραμματέας στην Σοβιετική Ένωση επενεύει και συνέβαλε όχι μόνο στην, στον αφοπλισμό αλλά και σε άλλα προγράμματα και από το 1985 ξεκίνησε η συνεργασία στην οποία βασίστηκε το πρόγραμμα ITER και δεν πρόκειται μόνο για μία απόφαση πολιτική αλλά για μία επιβεβαίωση ότι ο ψυχρός πόλεμος διεγράφηκε τελείως σε μία και διαπαντός και θέλω απλώς να σας πω ότι η σύνδεξη ε, ε, ε, οδήγησε το βραβείο Νόμπελ ενός Ούγγρου και εγώ σαν Ουγγαρέζα, σαν Ευρωπαία, σαν κάποιον που ζει σε αυτό το διεθνές περιβάλλον στηρίζω την προσπάθεια αυτή. Ε, θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε την πολιτική παραγωγή μόνο οικονομικά αλλά και ε, οικονομικά ε, για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριο Χάγκλουντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ειλικρινά Είμαι πολύ ικανοποιημένο με τον μόνιμο ε, εισηγητή για επιστημονικά θέματα και εκ μέρους της ομάδας μας. Ε, χαίρομαι που μπορέσαμε να βρούμε τρόπο να χρηματοδοτήσουμε πάλι το ΙΤΕΡ. Η όλη διαδικασία ήταν δύσκολη. Πρώτα απ' όλα κατέδειξε ότι το Συμβούλιο δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις τους και μάλιστα ούτε και στις πολιτικές του υποσχέσεις όσον αφορά την έρευνα. Ταυτόχρονα είδαμε μία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο ήθελε να μειώσει τα κονδύλια στο 1α που είναι ε, τα ερευνητικά προγράμματα. Εκεί χρηματοδοτούνται σχεδόν κατά 100% και υποστηρίζεται η στρατηγική του 2020. Θυμόσαστε η ιδέα ήταν να πάρουν τα χρήματα για την για το σχέδιο ίτερ από εδώ. Είπαμε όχι, ήμασταν ενωμένοι σαν κοινοβούλιο, ήταν σταθερή η θέση της Επιτροπής Προϋπολογισμού και τελικά καταλήξαμε σε θετικό αποτέλεσμα. Αλλά από την άποψη της ομάδας μας δεν είναι ιδανική η λύση. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Μελλοντικά συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Το σχέδιο Ίτερ έχει μεγάλο δυναμικό, είναι τεράστιο σχέδιο και ταυτόχρονα θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια έδειξαν ότι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ε, γνώση σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται το Ίτερ γιατί δίνουμε λεφτά των φορολογουμένων και κονδύλια και δεν πρέπει να υπάρχει τόσο κακή διαχείριση που να αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε σε τέτοιες λύσεις όπως η σημερινή για να σώσουμε το σχέδιο ΙΤΕΡ. Επίσης, στο επόμενο MFF θα πρέπει να έχουμε πιο σαφείς λύσεις για τη χρηματοδότηση, ώστε να μην βρισκόμαστε εδώ σε τρία χρόνια και σε πέντε χρόνια να επαναλαμβάνουμε τα ίδια όπως απόψε να μεταφέρουμε δηλαδή κονδύλια για να καλύψουμε τον προϋπολογισμό του σχεδίου ΙΤΕΡ. Θα ήθελα ακόμη να αναφέρω ότι το Συμβούλιο κοιμότανε. Μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία. Υπήρξαν ε, επαφές με στο Συμβούλιο. Κάποιες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο θέλαν να υπαναχωρήσουν ε, τελικά κατάλαβαν ότι δεν ήταν επιθυμητή μια τέτοια υπαναχώρηση και το Συμβούλιο θα μείνει σε αυτή τη συμφωνία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία, διότι ο ορίζοντας 2020 χρειάζεται όλα τα κονδύλια που μπορούμε να βρούμε. Πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε λύσεις μελλοντικά που να συνεπάγονται λιγότερα χρήματα, λιγότερα κονδύλια για ερευνητικά προγράμματα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Το αποτέλεσμα είναι καλό σε σχέση με τις συνθήκες. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Τζουνό, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είπατε ότι η κατάσταση δεν είναι ιδεώδης διότι η Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύω και για πολλά χρόνια ακόμη ε, φοβάμαι ότι αντιμετωπίζει κρίση, ε, δημοσιονομικά προβλήματα και όλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταρτήσουν και να ισοσκελίσουν τους προπολογισμού τους προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την Ευρώπη και τους πόρους της και τη στιγμή που ζητάμε να μειώσουμε τον προπολογισμό αποφασίζουμε αυτό που σκοπεύουμε να αποφασίσουμε τώρα. Είναι πράγματι πολύ δυσάρεστο διότι σήμερα και αύριο ζητούμε να επιβεβαιώσουμε τον διορθωτικό προϋπολογισμό για 650 επιπλέον ε, εκατομμύρια ευρώ για το 12 για το πρόγραμμα ITER και ε, να ε, υπάρξει 1,12% δισεκατομμύρια δηλαδή 1,2% του προϋπολογισμού της Ευρώπης ε, και διαθέτουμε αυτό το ποσό το οποίο ενδεχομένως το 2050 για τους πιο αισιόδεξου θα μπορέσει να τελεσφορήσει δηλαδή τρελαθήκαμε τελείως τη στιγμή που όλα πάνε κακά και προς το χειρότερο θέλουμε να διαθέσουμε αυτό το ποσό. Ίσως δεν μειώνουμε άλλους προϋπολογισμούς παρόλο που έχουμε περικόψει την Ευρώπη του 2020 και ούτω καθεξής αλλά ό,τι διατίθεται εδώ δεν διατίθεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας οι οποίες θα είχαν αμέσως αποτελέσματα όχι το 2050-2080 αλλά το 13-14 και θα δημιουργούσαν επιπλέον και θέσεις εργασίας. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε μία τέτοια τρέλα τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τόσες δυσκολίες. Κυρία Χέρτσοκ, μα θυμήσατε την ιστορία. Μας είπατε ότι ε, το πρόγραμμα αυτό καταρτίστηκε πριν 30 χρόνια, στο τέλος του ψυχρού πολέμου. Δεν πρέπει όμως να αναθεωρήσουμε τα προγράμματά δεν πρέπει ε, όταν οι Ευρωπαίοι φτωχαίνουν όταν δεν υπάρχουν προγράμματα όταν δεν ισοσκελίζονται οι προπολογισμοί και δεν μπορούμε εμείς να καταρτήσουμε προπολογισμό να διαθέσουμε 1,2 δισεκατομμύρια και εδώ δεν μιλάμε μόνο για το 12 αλλά μέχρι το 2020 θα συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη νομίζω ότι πραγματικά πρέπει κανείς να τρομάξει για αυτή την αρρωστημένη εξέλιξη τη στιγμή που όλα πάνε στραβά. Γι' αυτό και η πολιτική μου ομάδα δεν θα υπερψηφίσει αυτόν τον διορθωτικό προπολογισμό. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο για τρία λεπτά στον Ρίτσαρτ Άσφορντ. Αλλά βλέπω μία μπλε κάρτα για την κυρία Ντουρόν. Δέχεστε μία μπλε κάρτα κυρία Ντουρόν. Από την κυρία Χέρτσογκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Συζητάμε εδώ για τον ο, χάρτη πορείας της ενεργείας για το 2050 που δεν ανέρχεται στο 1985 σαν το ίτερ και αναρωτιέμαι αν οι πράσινοι θα στηρίξουν το χάρτη πορείας της ενεργείας για το 2050 διότι θα υπάρξουν αλλαγές μέσα στα επόμενα 35 χρόνια χρόνια. Κυρία Ντουρό, έχετε το λόγο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς βρισκόμαστε σε μια τεχνολογία του παρελθόντος. Το, η πυρηνική ενέργεια ανήκει στο παρελθόν και θα πρέπει να αλλάξουμε και ε, υπάρχει κάτι ιδεολογικό το οποίο, στο οποίο πιστεύουμε. Ορισμένοι λοιπόν πιστεύουν χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη ότι μέχρι το 2050 ή το 2080 θα έχουμε λύσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να εγκιστρωνόμαστε είμαστε έτσι και οι απαντήσεις οι οποίες μας έδωσαν οι μηχανικές δεν ήταν πιστικές και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζουμε να επιμένουμε σε αυτές τις ενέργειες του παρελθόντος. Και τώρα για τρία λεφτά ο κύριος Ρίτσαρντ Άσφορντ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον τομέα της έρευνας και για το λόγο αυτό σαφώς ε, υποστηρίζουμε το πρόγραμμα ITER. Για το λόγο αυτό θα υποστηρίξουμε και τη συμφωνία που πετεύθη με το Συμβούλιο. Καταλαβαίνουμε ότι θα σημαίνει επιπροσθέτως 350 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι μέρος του διορθωτικού προπολογισμού. Θα πρέπει να δηλώσω εδώ το ενδιαφέρον μου γιατί στην εκλογική μου περιφέρει ένα μεγάλο εργαστήριο στην Οξφόρδη. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εξασφαλίζοντας το μέλλον αυτού του εργαστηρίου θα εξασφαλίσουμε 500 θέσεις εργασίας ερευνητών, άτομα που βρίσκονται πολύ μπροστά στην τεχνολογία και αυτού του είδους ε, την εμπειρία δεν, δεν μπορούμε να, να χάσουμε. Θα ήθελα όμως να πω κάτι και να προειδοποιήσω. Η τεχνολογία εχμής πάρα πολύ συχνά κατηγορείται για αύξηση του κόστου. Έχοντα στο νου αυτό υπάρχουν τρία σημεία που θα ήθελα να τονίσω. Καταρχά, αυτή η επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να βρεθεί από τον υπάρχοντα προπολογισμό. Το 2012 δεν θα ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να παράσχουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Αυτό είναι απόλυτα σωστό γιατί οι κυβερνήσεις και οι προπολογισμοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλές πιέσεις. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και το 2013. Δεύτερον, Αυτά είναι χρήματα των φορολογουμένων. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει η πειθαρχία του προπολογισμού στην κοινότητα των ερευνητών. Είναι επίσης σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλουμε την προσεκτική, το προσεκτικό έλεγχο αυτής της βιομηχανίας. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε άμεση εμπλοκή. Κύριε Επιτροπή, Επίτροπε, θα να σας ζητήσω να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτό. Τέλος, για να διευκολύνουμε όλα τα παραπάνω, πιστεύω ότι είναι απόλυτα σημαντικό το πρόγραμμα ITER να ενταχθεί στο επόμενο επόμενο πολιετές ε, πλαίσιο ε, εδώ απαιτείται να υπάρχει, ε, να είμαστε υπόλογοι, απαιτείται να υπάρχει ένας προπολογισμός. Ευχαριστώ πολύ για δυόμιση λεπτά, κυρία Αντράσεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι κατά της σύνδεξης Παρ' όλα αυτά, όταν τίθεται το θέμα του ΙΤΕΡ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει μάθει από τα λάθη τη. Δυστυχώ δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Καλλιλέο, το οποίο κόστησε 700 εκατομμύρια ευρώ το 2000, το 2010 το υπολογισμένο κόστο τριπλασιάστηκε και συνεχίζει το κόστο αυτό να αναρριχάται. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικά όλα αυτά. Οι εταίροι μας ε, λένε ότι μπορεί να γίνει κάτι μέχρι το 2018, πέντε χρόνια αργότερα από την ημερομηνία που συμπεριλήφθη στην αρχική συμφωνία. Το πρώτο πίνα, τα πρώτα πειράμανα δεν ε, θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του 2025. Το κόστος ε, κατασκευής θα διπλασιαστεί από τους αρχικούς υπολογισμούς. Θα περάσουμε από τα 5 δις στα 10 δις. Το της λειτουργίας ε, Twitter ε, επιπλέον 5 δισεκατομμύρια και αυτό το κόστος θα αυξηθεί. Από τη στιγμή που το 90% του προγράμματος το διαχειρίζονται οι χώρες, οι συμμετέχουσες χώρες, δεν ξέρουμε, δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Νομίζω ότι οι, ε, οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το κόστος του ύστερα από τη στιγμή που το ε, πληρώνουν. Εδώ μιλάμε για την πρωτοδότηση ενός προγράμματος που κοστίζει 50% από τα προβλεπόμενα. νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή είναι καταστροφική. Ο Πίτροπο Λεμαντόφσκι μα είπε Δευτέρα ότι ο προβλεπισμό του 2011 ήταν επιπρόσθετο, ε, είχε επιπλέον ποσό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από μερικού μήνε μα είπε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα 11 εκατομμυρίων ευρώ. Με συγχωρείτε, τι από αυτά ισχύει. Δεν ξέρει πόσα χρήματα υπάρχουν ε, σήμερα. Εγώ το ξέρω και το ξέρουν και όλοι οι υπόλοιποι. Το ίτερο όπως και το πρόγραμμα Γαλιλαίο γίνεται μια, ένα, ένας παραλογισμός. αλλά οι ε, ε, πολίτες που καλούνται να, πληρώσουν γι' αυτό δεν ε, διασκεδάζουν καθόλου. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να απορριφθεί εντελώς αυτό το πρόγραμμα. μισή λεπτό τώρα ο κύριος Ράμακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι υπέρ ε, της πρόσθετης χρηματοδότησης του προγράμματος ίτερ για πολλούς λόγους. Εδώ και πολύ καιρό έχω την άποψη ότι η πυρηνική σύνδεξη θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για την ανθρωπότητα για να καλύψουμε ενεργειακές ελλείψεις. Υπάρχουν και άλλες βεβαίως εναλλακτικέ λύσεις ακόμη η Ευρώπη θα μπορέσει να προχωρήσει στην έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι που θέλουμε πάντα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα κονδύλια που έχουμε πρέπει να αφιερωθούν σε, ε, σε σχέδια κλειδιά με διαφανή τρόπο. Δεν θα πρέπει να διστάζουμε, πρέπει να βρίσκουμε χρήματα και κονδύλια για αυτά τα σημαντικά προγράμματα. Η κρίση δεν είναι επιχείρημα. Για να ξεπεράσουμε την κρίση χρειαζόμαστε σχέδια σαν το ΙΤΕΡ. Άλλωστε, το σχέδιο αυτό είναι μια ευκαιρία και για μικρότερα κράτη-μέλη και είναι και σημαντικό σχέδιο για τις μικρομεσαίες εταιρείες. 50% των συστατικών προέρχονται από ΜΜΕ. Θα είναι κρίμα να μην χρησιμοποιήσουμε τον ήλιο και το νερό προς όφελος της ανθρωπότητας, έστω και αν δεν ζούμε το για να δούμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Και τώρα προχωράμε στους επόμενους ομιλητής, ο κύριος Γκαρίγκα Πολέντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι που μείνατε τόσο αργά στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό. Πρέπει να πω ότι είναι ένα θαύμα που η Κομισιόν μπόρεσε με το Ευρωκοινοβούλιο να προχωρήσει. Θα ήθελα να συγχαρώ και τα δύο μέρη ε, διότι μπορέσαμε τέλος πάντων να βρούμε τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Εξάλλου αυτά τα 350 εκατομμύρια δεν έρχονται από μια ανακατανομή του 1α ένα μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από αναθεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε να επηρεάσουμε κάπως το Συμβούλιο και φροντίσαμε το Συμβούλιο να βάλει φρέσκα χρήματα για να ανταποκριθεί σε νέες χρηματοδοτικές ανάγκες, πράγμα το οποίο ανταποκρίνεται στις διεκδικήσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Διότι αν δεν επρόκειτο για νέα χρήματα δεν θα ήταν σωστή αυτή η δημοσιονομική πολιτική. Δεν είναι εύκολο βεβαίως να βρούμε 350 εκατομμύρια για το επόμενο χρόνο χωρίς να ζημιώσουμε προγράμματα που εξελίσσονται θα αντιμετωπίσουμε δυσχέρειες αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να προσπαθήσουμε ο προϋπολογισμός 2013 πρέπει να είναι επικοδομητικός δεν καταλαβαίνω ορισμένε πολιτικές ομάδες που χρησιμοποιούν σαν αιτιολόγηση την κρίση ε, ε, ο συνάδελφος το είπε μόλις πριν το πρόγραμμα ITER είναι πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Θα μας βοηθήσει να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία. Θα πρέπει να είμαστε οραματιστές. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε σε ορίζοντα 10 ετών ή 20 ετών. Είναι λάθος να θεωρήσουμε την κρίση σαν αιτιολόγηση αρνητική. Α ελπίσουμε ότι το Ήτρα θα μας δώσει νέα ενέργεια σε 10-20 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από την κυρία Ντυρόν. Κυρία Ντυρόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που δέχεστε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μου ε, ε, κάνει εντύπωση πώς παρουσιάζεται αυτό το πρόγραμμα σαν σημαντικό φάρο. Ε, ενώ κανένας μας δεν έχει τη βεβαιότητα ότι θα λύσει ε, ε, το, πρόβλημα, το πρόβλημα το ανεργειακό και δεν είναι άλλοθη η κρίση. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι, είναι ο προσδιορισμός οποιοδήποτε προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο πρόγραμμα 2020 όπως το προβλέπουμε και βεβαίως δεν μπορώ να δεχθώ αυτό που είπατε ότι είναι άλλοθη η κρίση. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κυρία Ντουράν. Κοιτάξτε, μία εκπρόσωπος των Πρασίνων να μου λέει ότι πρέπει να έχω επαφή με την πραγματικότητα. Με εκπλήσει γιατί είναι μέρος του πολιτικού σας προγράμματος η αναζήτηση νέων εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Αυτή είναι μία εναλλακτική μορφή. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για την ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη κάθε περίπτωση με την, με την τεχνολογική στήριξη που δίνεται σε αυτό το πρόγραμμα νομίζω το 1,3 εκατομμύρια δεν είναι και πάρα πολλά χρήματα. Ο κύριος Τικάο για δύο λεπτά. Κυ... Κύριε Πρόεδρε, Το πρόγραμμα αυτό μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε καθαρή ενέργεια η πειραματική φάση του ΙΤΕΡ και του, της σύνδεξης και του πυρηνικού σταθμού που ετοιμάζεται στη Γαλλία ετοιμάζει τη νέα γενιά των αντιδραστήρων και θα βοηθήσει την Ευρώπη να περάσει ακριβώς σε αυτούς τους πειραματικούς και οριστικούς αντιδραστήρες. Η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου του 2011 δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις δαπάνες του ΙΤΕΡ για το 2012 μέχρι 2015. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια μπαίνουν στον προϋπολογισμό του 12, 360 θα είναι πιστώσεις για το 13 και τα κατόφλι για το 1α θα αυξηθεί κατά 840 εκατομμύρια. και έχουμε 190 στο 2013. Αυτά είναι η αύξηση στον τομέα 1α νότου το όριο PDP. Λοιπόν, υποστηρίζω το πρόγραμμα ITER. Το ποσό των 650 είναι πρόσθετο. Έτσι όμως τηρείται και η συμφωνία που υπογράφηκε. Ένα λεπτό, ο κύριος Ενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια έρευνας για να μπορέσει να υπάρξει διεθνής συνεργασία η οποία να προσβλέπει προς το μέλλον. Με την θερμοπυρηνική σύνδεξη θα υπάρξει μία ενέργεια που δεν θα ρηπαίνει, θα είναι προσβάσιμη σε όλους και δεν θα κοστίζει πολύ. Και η η επιτυχία του ΙΤΕΡ είναι πολύ σημαντική διότι θα αυξηθούν οι ενεργειακές μας ανάγκες και δεν μπορούμε να γυρίσουμε ε, την ε, πλάτη της ε, τις επιθέσεις του τομέα της ενέργειας διότι θα πρέπει να δημιουργηθούν δημόσιες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα που θα απαντήσουν στις προκλήσεις που παρουσιάζει το ΙΤΕΡ να έχουμε μια οικολογική, έναν οικολογικό προγραμματισμό για τις μεταφορές, για την διανομή και για να μην υπάρξουν μεγάλα ατυχήματα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Χολμάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Για το ΊΤΕΡ μιλάμε για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα έρευνας, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι σε κάθε κρίση και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε θα εγκαταλείπουμε την έρευνα και τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε ε, συνάψει και δεν θα τις σεβόμαστε πλέον. Πρέπει να ε, υπάρξει μία ε, τεχνολογία του μέλλοντος και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο με έχει προβληματίσει διότι βλέπω ότι δεν προχώρησε παρκώς το πρόγραμμα αυτό διότι στην αρχή δεν είχαμε τη δυνατότητα των υπολογιστών την οποία διαθέτουμε τώρα και δεν είχαμε τα υλικά τα οποία απαιτούνται για τις υψηλές θερμοκρασίες εξού και μέχρι στιγμής η έρευνα δεν προχώρησε ομαλά στο θέμα του ίτερ. Χρειάζεται όμως για τα μεγάλα προγράμματα να υπάρχει από την αρχή μία σωστή ε, χρηματική στήριξη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει ε, σε πολλούς τομείς ε, τότε θα πρέπει από την αρχή τα προγράμματα αυτά να έχουν μία επαγγελματική διαχείριση των προγραμμάτων ε, να γίνει ένας σωστός και ρεαλιστικός υπολογισμός του κόστους και όχι μόνο μία πολιτική ωρεοποίηση των στοιχείων και να υπάρξει εποπτεία και παρακολούθηση κατά τρόπον ώστε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πάντοτε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται τα έξοδα διότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που θα κρατήσει κρατήσει χρόνια. Γι' αυτό και είναι σημαντικό εφόσον και εγώ είχα πάει στο Κανταράς και είδα τις εγκαταστάσεις όπως και εσείς κυρία Ντουρό θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το πρόγραμμα και να θεωρήσουμε ότι είναι μια προοδική για το μέλλον. Ευχαριστώ. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Φρονκό. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπο και κύριοι συνάδελφοι. Χαίρομαι που αυτός ο διορθωτικός προπολογισμό που αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ και που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Προπολογισμού στις 29 Μαρτίου, χρηματοδοτώντας αυτό το επιπλέον κόστος, Αποφεύγουμε το να πετάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο έρευνα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει καθοριστικό ρόλο και βεβαίω τιμάμε τι συμφωνίες, τις διεθνείς συμφωνίες. θα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι κανένα από του 7 εταίρου τη Επιτροπή Euratom δεν αμφισβήτησε τη συνολική του συμβολή στο πρόγραμμα αυτό η Ιαπωνία παρόλο το δράμα τη Φουκουσίμα αποφάσισε να σεβαστεί κατά γράμμα τις υποχρεώσεις του προπολογισμού σε ό,τι αφορά το ΙΤΕΡ. Δίχως αυτή τη συμφωνία πάρα πολλοί ερευνητέ θα πρέπει να σταματήσουν να, να, να, εργάζονται και θα υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις. Σήμερα ένα εκατομμύριο άτομα εργάζονται ε, για το ΙΤΕΡ στο Καταράζ. Ε, ε, το 2018 ε, θα μπορούσαν να, να, να αυτό θα, μπορούσαν να δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Συμπερασματικά κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είμαστε περήφανοι και είναι σύμβολο αριστείας για την Ευρώπη το ΙΤΕΡ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με τους ομιλητές και μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συνδιαδικασία Catch Έχω μόνο μία έτοιμα αγόρευση της κυρίας Πασεκού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή είναι μια διοργανική συμφωνία και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα να μπορέσει να περατωθεί και η συμφωνία που πετεύχθη είναι προς το συμφέρον μας. Το ΙΤΕΡ θα είναι δίχως άλλο ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των άλλων θα μπορούσε να προετοιμάσει το δρόμο για μια ασφαλή πηγή ανέργειας χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Συμφωνώ με τη μακροπρόθεσμη εγγύηση χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγγυηθεί την επιτυχία του προγράμματος σε ένα αποδεκτό κόστος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς δεσμεύσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, ουσιαστικά πρόκειται για ένα διυπηρετικό πρόγραμμα το οποίο πρόκειται ε, να προσφέρει ε, κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και είναι θέμα αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια υπάρχουν υπερβάσεις κόστους και ένα πρόβλημα διαχειριστικό το οποίο οφείλεται εις την κοινή προσπάθεια για την σύνδεξη αλλά είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο και υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγής. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την υπέρβαση κόστους αυτού του διπυρωτικού προγράμματος και θέλω να πω και στην κυρία Σεν σχετικά με τη λογική του προϋπολογισμού του 2011 το οποίο υπέφερε διότι είχαμε 10 ε, εκατομμύρια τα οποία δεν είχαν καταβληθεί για νόμιμα προγράμματα πρώτον διότι δεν υπήρχε ε, ευελιξία στον δημοσιονομικό κανονισμό και δεν είχαμε επάρκεια πόρων. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε τώρα να επιλύσουμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε επιπρόσθετα έσοδα για τον προπολογισμό του 2012 για να αποφύγουμε ε, τα, ε, τα ε, ε, ελλείμματα και να έχουμε πλεονάσματα και να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτά που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί το 2011. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Μπαλτζάνη για να καταλήξει. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμερίστηκαν μαζί μου αυτή την έκθεση που συζητάμε. Θα ήθελα να πω στην συζήτηση αντιμετωπίσαμε το θέμα, την ουσία αυτού του προγράμματος ίτερ. Θα ήθελα όμως να θυμίσω ότι σήμερα πραγματικά εφαρμόζουμε τη συμφωνία που προσυπεγράφει το Δεκέμβριο και που μας επέτρεψε να περατώσουμε τη συμφωνία για τον προπολογισμό του 2012. Εφαρμόζουμε δηλαδή ε, μια συμφωνία που έγινε στα πλαίσια της συνδιαλλαγής που σηματοδότησε το πέρας της, ε, το συζητήριο του προπολογισμού και μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε αυτόν τον καλύτερο δυνατό κόσμο. Γιατί για να χρηματοδοτηθεί το σημαντικό αυτό πρόγραμμα χρησιμοποιούμε στο, ε, στο ελάχιστο το μέσο των υπολείπων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν διακυβεύονται τα άλλα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται με βάση τον προπολογισμό. Συνεπώς αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Και πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή η συνδιαλλαγή αποτέλεσε το, την τελευταία φάση διαπραγματεύσεων που έγιναν σε πνεύμα συνεργασίας που ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. The debate is just now finished and... Έληξε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση